Το πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής και η αποτελεσματικότητά τους. Θα γίνει παρουσίαση της μελέτης και ανταλλαγή απόψεων. Η κυρία Χόλμαγερ, η δυστυχώ δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρούσα στη συνάντηση σήμερα. Ζήτησε από τον Μάρκους Πίπερ να την εκπροσωπήσει. Ο Μάρκους θα έχει το λόγο λοιπόν για την γνωμοδότηση Χολμάγερος προς το περιεχόμενο της μελέτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μελέτη αξιολογήθηκε από την κυρία Χολμαέρ με τα εξής αποτελέσματα. Το ένα είναι πως Το ένα ήταν η εξολόγηση που έγινε από το τμήμα πολιτικής εδώ πέρα. Για το εάν η προώθηση και η οι επιδοτήσεις ε, των ε, επενδύσεων ε, έχουν προβλήματα με τους φακέλους. Γνωρίζετε πως έχουμε κάποια ζητήματα γιατί ξέρετε πως υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να δημιουργηθούν χι θέσεις εργασίας, αν, πρέπει, αν υπάρχει μια συγκεκριμένος βαθμός καινοτομίας και μετά πρέπει να αποδείξει κανείς, να υποβάλει τα δικαιολογικά για να αποδείξει ότι τα έκανε αυτά τα πράγματα και είναι από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ, πάρα πολύ ε, περίπλοκο. Και υπάρχουν κάποιες ε, κατευθυντήρες γραμμές, κάποιοι δείκτες ε, ε, με τους οποίους μπορούμε απλούστερα να μετρήσουμε την κατάσταση. Και θεωρώ πως πως ε, όταν μιλάμε για διαρθρωτικά ταμεία μπορούμε κάπως να βελτιώσουμε την ε, κατάσταση. Βέβαια το θέμα είναι τι θέλουμε να επιτύχουμε με αυτά τα κονδύλια. Αυτό το οποίο βρίσκω εγώ πολύ ενδιαφέρον είναι μια αξιολόγηση της ε, λογικής ε, εκθεμελίων αξιολόγηση της λογικής των επιδοτήσεων για αυτό το αντικείμενο, γιατί συχνά ε, καταλήγουν αυτά τα πράγματα σε μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν ούτως ή άλλως και απλά εντάξει μετά έχουν και κάποια άλλα έσοδα κατά το οποίο είναι ευχάριστο αλλά δεν είναι καθοριστικό. Και βεβαίω αυτή η αλλως και απλα ενταξει μετα εχουν και καποια αλλα εσοδα κατα το οποιο ειναι ευχαριστο αλλα δεν ειναι καθοριστικο και βεβαιως αυτη η εμπειρια θα παρατηρείτε και σε πολλά σημεία της ε, Ευρώπης. Δηλαδή κάποιες εταιρείες εγκαθίστανται κάπου λόγω των συγκοινωνιακών συνδέσεων, λόγω της τιμής ενέργειας και οπωσδήποτε λόγω των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Και επιβεβαιώσαμε αυτό το οποίο έλεγε η Κομισιόν. Λυπηρό βρίσκω το ότι ε, δυστυχώς είχε αντίθετη άποψη ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, περιφερειακών θεμάτων γιατί ήθελε να μπορούν ακόμα να παίρνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις επιδοτήσεις στις περιφέρειες. Κάτι το οποίο είναι αντίθετο με τα ευρήματα αυτής της ε, μελέτης. Θα το δούμε βεβαίως. Απλά σα λέω πού πάνε και οι διαπραγματεύσεις του τριμερούς ε, διαλόγου. Γιατί πρέπει να έχουμε βεβαίως πάντα κατά νου τις ε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές θέλουμε να στηρίξουμε. Αυτά έτσι ως κάποια πρώτα αποτελέσματα της μελέτης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να καλωσορίσουμε τους συντάκτες της έκθεσης και θα τους δώσουμε το λόγο για 15-20 λεπτά ώστε να έχουμε τα βασικά στοιχεία της έκθεσης. Και για να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων και ένας γύρος συζητήσεων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για την εισαγωγή, κύριε Πίπερ. Πραγματικά μπήκατε σε ένα από τα βασικά μηνύματα της μελέτης. Και η βιβλιογραφική έρευνα που έχουμε κάνει δείχνει ότι όταν μια επιχείρηση αποφασίζει να μετακινηθεί σε συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να είναι ελκυστικά τα κονδύλια από την Ένωση αλλά δεν είναι αποφασιστικός παράγοντας. Άλλοι παράγοντες ε, ε, παίζουν οι εγκύτες στην αγορά, μεταφορές, η βιβλιογραφία δείχνει ότι αυτοί είναι οι καθοριστικοί παράγοντες. Να σας παρουσιάσω τη μελέτη εντάχει. Δεν γίνεται το τελευταίο εξάμεινο. Και θα σας πω και δύο λόγια για τους στόχους και τη μέθοδο. Περιγράφοντας κατόπιν και τα κύρια ευρήματα. Στόχοι. Τι θέλει να πετύχει η μελέτη. Δύο βασικά θέματα. Τις κανονιστικές απαιτήσεις, αυτές που αποκαλούνται ε, απαιτήσει ε, διάρκειας του άρθρου 57. Το τι λέει το άρθρο αυτό είναι κάπως περίπλοκο θέμα. Απαιτεί ο δικαιούχος των διαθωτικών πόρων, κάποιος που έλαβε κάποιο κονδύλι και το επένδυσε σε μια παραγωγική επένδυση, να κρατήσει την επένδυση αυτή για πέντε χρόνια τουλάχιστον μετά την ολοκλήρωση της δράσης. Υπάρχουν εξαιρέσεις, μπορεί να γίνει τρία χρόνια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι άλλες εξαιρέσεις που σταδιακά εντάσσονται στις απαιτήσει ε, διάρκειας. Κάτι άλλο σημαντικό στο 57 αφορά την επανεγκατάσταση. Το άρθρο 57 προβλέπει ότι μια επιχείρηση που έχει πάρει μέτρο αποκατάσταση το μέτρο επιστροφής γιατί μετακινήθηκε αλλού δεν μπορεί να πάρει κονδύλια, άλλα κονδύλια από τα διαθροτικά ταμεία. Πέραν της διάρκειας η διάρκεια είναι σημαντικός ε, παράγοντας ε, στα διαθροντικά ταμεία. Είναι γύρω στα 70, δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά, εκ των οποίων ένα μεγάλο ποσοστό είναι βιώσιμο. Και το, η έννοια βιωσιμότητα δεν είναι, ε, σημαίνει σε εμάς δυνατότητα διάρκειας μετά το πέρας της ε, περίοδου υποστήριξης. Το γράφημα σας δείχνει την κατανομή γενικά των 70 δις. 40% περίπου πηγαίνουν σε άμεση ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ένα άλλο 40% υποστήριξη σε μεγάλες επιχειρήσεις και 20% αναδιάρθρωση και προσαρμογή των εργαζομένων βάσει του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Τώρα, γιατί πρέπει να ανησυχούμε για τη διάρκεια, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Στην παρουσίαση του, της θεματικής υποστήριξης επιχειρήσεων η Επιτροπή έδωσε κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Το 50% των επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν στην Ένωση μόνο το 50% επιβίωσε την πρώτη πενταετία. Εδώ βλέπετε τις λεπτομέρειες των επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν το 2008, πόσες υπάρχουν ακόμα δύο χρόνια μετά, το 2010. Όπως βλέπετε υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Κάποιες χώρες έχουν καλή βιωσιμότητα πάνω από 80%, σε άλλες τα νούμερα είναι μικρότερα. Ε, η μετακίνηση επιχειρήσεων ήταν μεγάλη ανησυχία στο Κοινοβούλιο. Εμείς εξετάσαμε τα ερωτήματα του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό την τελευταία περίοδο και βρήκαμε καμιά κατοστή ερωτήσεις για θέματα μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. Είναι συνήθως ευρωβουλευτές που ανησυχούν γιατί μία επιχείρηση στην περιοχή τους πήγε κάπου αλλού στην Ένωση και πήρε χρηματοδότηση της Ένωσης σε κάποια φάση. Τα νούμερα, βλέπετε τα νούμερα εδώ που δείχνουν από ποιους προήλθαν οι ερωτήσεις. 19 από το Γάλλοι βουλευτές που έδειξαν ησυχία για τη μετακίνηση μιας επιχειρήσης μεγάλη συνήθως κάπου αλλού και ρωτούν αν πήρε κονδύλια κάποια στιγμή στην ιστορία της από την Ένωση. Πώς έγινε αυτό. Μελετήσαμε την κατάσταση, όχι μόνο με τα εφιστάμενα αλλά και με τα παρελθόντα νομοθετικά κείμενα των διευθυντικών ταμείων και με, είχαμε και άτομα, όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Πίπερ, έγινε μια σημαντική αλλαγή. Η διάρθρωση των απαιτήσεων βιωσιμότητας για την περίοδο 14 20 προβλέπει την ε, εξαίρεση των μεγάλων ενισχύσεων των άμεσων ενισχύσεων στις μεγάλες επιχειρήσεις. Συζητήσαμε και με τους διευθυντές των εποπτικών αρχών διαθωτικών ταμείων επιτόπου που είχαν μεγάλη εμπειρία μιλήσαμε με 67 διαχειριστικές αρχές και 42 ελεγκτικές αρχές, ενώ πήγαμε και επί τόπου, μιλήσαμε και με κάποιες από αυτές για θέματα βιωσιμότητας και διάρκειας. Τώρα, ποια είναι τα κύρια ευρήματά μας. Η ε, δική μας εξέταση του κανονιστικού πλαισίου ε, διαπιστώνει ότι υπάρχει σωστή αδιάρθρωση το, της βιωσιμότητας στα βιωτικά ταμεία και αυτό βελτιώνεται. Με το σχέδιο του νέου κανονισμού υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην βιωσιμότητα. Και οι απαιτήσει διάρκεια, η διάρθρωση και ο σχεδιασμό των απαιτήσεων αυτών βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έγινε πιο, πιο επακριβής, πιο λεπτομερής, ενώ λαμβάνονται υπόψη και η κρίση και δημιουργούνται εξαιρέσεις. Δηλαδή, αν ας πούμε δεν υπάρχει ευθύνη του ιδιοκτήτη για την διακοπή λειτουργία δεν απαιτείται η επιστροφή. Μιλήσαμε τώρα και με τους εμπλεκόμενους, τόσο τις διαφορετικές αρχές όσο και τους δικαιούχους των διαφορετικών πόρων. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανησυχία γιατί φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να, εφαρμοστεί, να εφαρμοστούν οι απαιτήσει του άρθρου 57 της Ένωσης. Βλέπουμε ότι τα κύρια προβλήματα είναι και πληροφόρηση αλλά και πολιτικά εμπόδια. Μια παραγωγική δραστηριότητα πρέπει να διατηρηθεί για πέντε χρόνια, δεν πρέπει να υπάρξει σημαντική, οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή τη δράση ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αυτό δεν είναι εύκολο να επαληθευτεί πάντα από τους ελεγκτές μας, ιδίως στις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πολύ δύσκολο πλαίσιο επιχειρηματικής λειτουργίας και είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσεις τι μεταβιβάστηκε, τι διαφυλάχθηκε και προφανώς οι επιχειρήσεις που ελέγχονται δεν τα λένε ξεκάθαρα τα πράγματα, ούτε δίνουν πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχει και ένα caveat, μια προσοχή, ένα σημείο προσοχής. Και στην όλη μελέτη, όπως ξέρετε, άρχισε κάπως να ξεκινήσει η περίοδος ε, των διαφορετικών ταμείων. Κάποια από αυτά άρχισαν να λειτουργούν το 8 ή το 9 και η πενταετία για αυτούς ξεκινάει πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της δράσης. Ε, ή τώρα στην πράξη. Τώρα του χρόνου αν αρχίσει λοιπόν να εξετάζει κανείς τις αιτήσεις εκθέσεις τις εκθέσεις συμμόρφωσης με το 57 δεν είναι πλήρης η εικόνα γιατί δεν έχουν ολοποιηθεί όλες οι... όλοι οι έλεγχοι. Να σας δώσω και κάποια στοιχεία από τις διαχειριστικές αρχές. Κάπου 80% θεωρούν ότι το άρθρο είναι σαφές, αρκετά σαφές. Η εικόνα αλλάζει σημαντικά όταν έχουμε την άποψη των επιχειρήσεων. Εδώ 40% περίπου από αυτούς που ρωτήθηκαν θεωρούν ότι το νοκανονιστικό πλαίσιο είναι ανεπαρκώς σαφές. Υπάρχουν καθηγητήρες γραμμές και από την και τα κρατη και υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της, ε, των καθηγητήριων γραμμών. Τώρα, ποια είναι τα προβλήματα των διαχειριστικών αρχών. Οι πληροφορίες που έχουμε μας λένε ότι είναι, οι αμφιβολίες σχετίζονται με τον σύνθετο χαρακτήρα των επιχειρησιακών δομών. 52% ε, η εταιρική νομοθεσία δεν είναι τόσο προβληματική, αλλά 52% συνεχίζουν να πιστεύουν ότι ε, και αυτό επηρεάζει. Πάντως ε, μια μεγάλη πλειοψηφία πάνω από 60% των αρχών θεωρούν ότι το άρθρο 57 είναι αποτελεσματικό. Η μελέτη επίσης ε, επικοινώνησε απευθείας με τις επιχειρήσεις που έλαβαν υποστήριξη για να τις ρωτήσουν τι συνέβαλε στη διάρκεια και τη βιωσιμότητά τους ε, οι κύριοι δείκτες βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις έχουν να κάνουν είτε με το σχεδιασμό της ε, δράσης ή την υλοποίηση και τα κριτήρια καθώς και το, οικονομικό, το χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Επιχειρήσεις για παράδειγμα που έχουν ε, ισχυρά θεματική, ισχυρή θεματική έμφαση με υποστήριξη από σωστό business plan, καλή εταιρεία, καλ, καλά partnership, αυτά βοηθούν την βιωσιμότητα. Αντίστοιχη εμπειρία είναι και η προσέγγιση των αρμο... η εγκύτητα μάλλον με τις αρμόδιες αρχές. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα από αυτά που μας είπαν. Θα κλείσω με κάποιες συστάσεις. Αυτό που σαφώς προήλθε από την εξέταση που κάναμε είναι ότι μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω την ε, καθοδήγηση για το πώς θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος της συμμόρφωσης με το μελλοντικό άρθρο 61. Για παράδειγμα, θα βοηθούσαν ίσως μελέτες περιπτώσεων και studies. Ή θα βοηθούσε αν ε, ερχόντουσαν οι αρχές, οι αρμόδιες αρχές και εξηγούσαν τι σημαίνει κάθε μέτρο. Επίσης, πιστεύουμε ότι θα ήταν καλό να υπάρχει περισσότερη διάδοση. Αρκετές αρχές ε, διαχειριστικές χρησιμοποιούν δείκτες για να δείχνουν τι πρέπει να πετύχουν, αλλού ωστόσο δεν έχει χρησιμοποιηθεί η, η διάσταση της διάδοσης επαρκώς. Δεν υπάρχουν δηλαδή καθοδηγητήρες γραμμές για το πώς ακριβώς θα μετράτε η συμμόρφωση με το 57. Επίσης είδαμε τη μεγάλη προσπάθεια αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής προγραμματισμού. Ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε πιο προσεκτικά και πιο λεπτομεριακά το θέμα του business support που δεν έχει και πολύ δουλειά και να έχουμε κάποιες πληροφορίες. Θα ήταν μια σημαντική συνεισφορά αν στο, πρόγραμμα, στο πλαίσιο των ελέγχων του το ελεγκτικό συνέδριο έθετε και το ζήτημα της βιωσιμότητας. Το κάνει ένα διαστήματα, αλλά συνολικά τα θέματα είναι... Το θέμα είναι κυρίως για αυτούς η αποτελεσματικότητα, όχι η βιωσιμότητα. Και τέλος θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διάδοση, αλλά διάδοση to the point, δηλαδή εξειδικευμένη διάδοση. Εξετάσαμε πολλά δεδομένα βέλτιστων ή καλών πρακτικών που υπάρχουν ήδη Πολλά μπορεί να γίνουν. Η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων έχει μια βάση δεδομένων σχετικά και περί τις 900 περιπτώσεις υποστηρίζονται από, τα, από κονδύλια της Ένωσης χωρίς να υπάρχει πουθενά μενία για την βιωσιμότητα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο γιατί σε μερικές περιπτώσεις δεν εμφανίστε παρκώς. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις. Eh, Να είστε καλά. Κύριε Μπλόμαγερ, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίασή σας. Κυρίες και κύριοι, Ας προχωρήσουμε στο, στην ανταλλαγή των απόψεων. Ποιος θέλει το λόγο? Θέλει να υποβάλλετε ερωτήσεις ή να μιλήσετε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω εξ αρχής ότι Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος ε, Πίπερ στην αρχή ξενόματος της ηγετρίας. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτό όμως που θέλω να υπογραμμίσω ε, είναι δύο λέξεις, durability και effectiveness, ε, διάρκεια και αποτελεσματικότητα οι πληροφορίες που είχαμε για την μη βιωσιμότητα ε, επιχειρήσεων που χρησιμοποίησαν τα χρήματα αυτά ε, μας δείχνουν ότι είναι ασθενής ε, η διάρκεια. 69 δις ευρώ έχουν δοθεί και ε, που δημιούργησαν θέσει εργασία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παρέμειναν οι ενδιαφερόμενοι στην εργασία. Ε, βλέπουμε ενδεχομένως και ε, αύξηση του εισοδήματος, αλλά και αυτό δεν έχει διάρκεια. Δηλαδή εδώ μιλάμε μονάχα για χρήματα τα οποία δαπανώνται ένομα σύμφωνα με τα όσα προβλέπει τον κανονισμό ή μήπω πρέπει να μιλάμε για την καλή αποτελεσματική χρήση των χρημάτων έτσι ώστε να υπάρχει πραγματική αποτελεσματικότητα γιατί φοβούμε ότι όλη αυτή η δομή στην οποία, στην οποία συμμετέχει και η Κομισιόν και οι τοπικές αρχές και οι εθνικές αρχές κτλ χρησιμοποιούν, δαπανούν τα χρήματα ε, χωρίς ε, όμως να προσπαθούν ε, να κάνουν επενδύσεις οι οποίες θα, από τις οποίες θα προκύψει επιστροφή των χρημάτων. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια λέμε. Υπάρχει φαίνεται μια νέα βιομηχανία στις χώρες στις δικαιούχες χώρες και βλέπουμε ότι είτε κανείς ε, ε, ότι για projects τα οποία μπορεί να κοστίζουν ε, είτε 5.000 είτε 50 εκατομμύρια το κόστος για την ίδια την μελέτη είναι το 10% ας πούμε του προϋπολογισμού. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για βιωσιμότητα, αλλά ποιος θα την προωθήσει και ποιος θα, την θα... υποχρεώσει τους ενδιαφερόμενους, οι τοπικές αρχές, οι ευρωπαϊκές και οι δύο. Ε, είπατε ε, ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο ε, να καθορίσουμε την αηφορία. Επίσης, η η οικονομική κρίση ε, έχει αλλάξει όχι μονάχα τα οικονομικά δεδομένα, αλλά ενδεχομένω και τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές ε, αρχές αντιμετωπίζουν ε, τα δεδομένα. Δηλαδή, τι πρέπει να καταλάβουμε, ότι θα πρέπει τα κονδύλια να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις προτεραιότητες τις οποίες καταρτίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς ή το ιδιωτικό τομέα ή μήπως θα πρέπει να υπάρξουν πιο όρημα ε, προγράμματα τα οποία θα λάβει υπόψη της ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της προστιθέμενης ευρωπαϊκής αξίας που μπορούν ε, να δώσουν Δηλαδή μπορεί να δοθεί μια όθηση έτσι ώστε να μειωθούν τα χάσματα ε, γιατί ε, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα προβληματικές καταστάσεις αλλά εγώ συγκεκριμένα στοιχεία από αυτού δεν βρίσκω σε αυτή την έκθεση. Κατά την άποψή σας, σε αυτή τη μελέτη μάλλον, η φυσική γυτνίαση ανάμεσα στους δικαιούχους και τις αρχές που διαχειρίζονται τα διευθυντικά ταμεία. Αυτό το αναφέρεται. Αλλά ποιος είναι πιο πολύ υπεύθυνο ε, για τα οικονομικά. Μπορού, πώς μπορούμε να ε, χωρίσουμε τις αρμοδιότητες, ε, πώς μπορούμε να τους χωρίσουμε ή μπορούμε, πώς μπορούμε να τους φέρουμε πιο κοντά. You gave Παραδείγματα ενδεχομένως. Έχω την αίσθηση ότι μπορούν να υπάρχουν ε, ε, παραδείγματα καλών πρακτικών αλλά που αφορούν μονάχα αυτό το 50% που έχουν ε, καταφέρει να νικήσουν το χρόνο και να έχουν διάρκεια. Επίσης, ποιος είναι ο ρόλος του ελεγκτικού συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. λέγεται ότι αναφέρεται στη σελίδα 69 ότι δεν, ε, έχει, δεν σχετίζεται με την ε, αηφορία ε, η οικονομική διαχείριση και επίσης λέτε ότι το νομοθετικό πλαίσιο για το 2000, για την επταετία 14 ή 20 θα πρέπει να ε, ε, ληφθεί υπόψη με διαφορετικό ε, τρόπο και όχι μονάχα από την, από την πλευρά του οικονομικού ελέγχου. Είναι σωστό αυτό ή γιατί εγώ διακρίνω μια αντίφαση. Επίσης, από τη μία πλευρά έχουμε τους γενικούς κανόνες της Κομισιόν και από την άλλη έχουμε τους ε, κανόνες που ε, εισάγονται από τις εσωτερικές αρμόδιες αρχές, ξεκινώντας από την ε, πολωνική εμπειρία και μη λησμονείται ότι είναι μεγάλη δικαιούχος η Πολωνία φοβούμε ότι αυτή η αρχική δημιουργικότητα τελικά είναι κακή για το project όταν ε, ακολουθούνται από πολύ κοντά ε, οι συμβουλές, οι αρχές και οι κανονισμοί. Εν πάση περιπτώσει, γενικά μπορώ να πω ότι η, μελέτη μάλλον είναι καλή. Μας δώσατε ε, στοιχεία συγκεκριμένα, μας δώσατε και την δυνατότητα να καταλάβουμε ε, ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε ένα καλό ε, πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σωστά. Αλλά αυτά είναι τα λόγια. Κύριε Μπλουμέγερ, θα πρέπει να είσαστε πιο θαραλέους και να ε, προσπαθήσετε να απαντήσετε χωρίς διπλωματία, δηλαδή με ένα ναι ή με ένα όχι, με ένα είναι θετικό ή είναι αρνητικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και αυτούς που έκαναν την παρουσίαση. Το πρώτο θέμα το οποίο ήθελα να πω είναι η απλοποίηση για να είναι αποτελεσματικότερη η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Γιατί ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει πρώτα να κάνουν αίτηση και μετά να εκταμιεύσουν και βέβαια θεωρούν πως είναι δύσκολη και γραφειοκρατική η διαδικασία. Έχετε κάποια άποψη λοιπόν για το πώς μπορεί να γίνει το σύστημα πλούστερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι ζήτημα όχι μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για οποιοδήποτε έργο του, ιδιωτικού, του εθελοντικού τομέα, των τοπικών αρχών, που συχνά ζητάνε ευρωπαϊκά κονδύλια, λαμβάνουν τη χρηματοδότηση και όταν τελειώσει η χρηματοδότηση σταματάει το έργο. Γιατί υπάρχουν προβλήματα βιωσιμότητας. Αναφέρατε το ζήτημα των βέλτιστων πρακτικών. Θα μπορούσατε νομίζω να μας δώσετε κάποια παραδείγματα, εάν υπάρχουν. Το άλλο αφορά την αιρεσιμότητα. Και, να αρχίσουμε εάν έχει ζητηθεί από κανέναν φορέα ο οποίος κάνει έτσι να επιδείξει ότι έχει σκεφτεί την ε, βιωσιμότητα του πρόγραμματος. Μάλιστα δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητάει το λόγο. Γι' αυτό θα δώσω λόγο στον κύριο Μπλωμαϊά. Μπορεί να απαντήσει. Και μετά ο κύριος Ιλαντ της Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί. Ευχαριστώ. Αν θέλετε με το υλικό που μας δίνετε μπορεί να κάνουμε μια άλλη μελέτη. Εγώ προσπάθησα να σας απαντήσω. Κάποια θέματα δεν τα είδαμε. Είναι εδώ και εκπρόσωποι της Επιτροπής. Δεν ξέρω αν είναι και από το Ελληνικό Συνέδριο που μπορούν να δώσουν τη δική τους άποψη. Για το πρώτο σας σχόλιο, τη σχέση μεταξύ αποτελεσματικότητας και διάρκειας και γιατί υπάρχει αυτή η απέτηση. Μπορώ να σας πω τι μας είπαν οι επιχειρήσεις. Θέλουν ευελιξία. Δηλαδή η απέτηση διάρκειας για αυτούς δεν έχει νόημα. Φερρυπίν, ας σκεφτούμε ένα έργο που επένδυσε σε software, σε λογισμικό και από, μετά από 2-3 χρόνια δεν είναι χρήσιμο το λογισμικό. Θα πρέπει να ξεκινήσουν να επενδύουν σε κάτι καινούριο, ενημερωμένο λογισμικό. Το να τους το επιβάλλουμε να το κρατήσουν δεν έχει νόημα. Όταν μελετούσαμε τις τροπολογίες που είχε υποβάλει το Κοινοβούλιο στις προτάσεις επιτροπής για το νέο γενικό κανονισμό υπήρχαν κάποια σημεία που ζητούσαν να επανεξεταστεί η πενταετία ή τριετία σε περίπτωση τεχνολογικής έρευνας, όταν οι τεχνολογικές αλλαγές εξελίσσονταν ταχύτερα. Και υπάρχουν και οι πληροφορίες που πήραμε από τις επιχειρήσεις που είπαν ότι σε κάποιες περιπτώσεις η απέτηση πενταετίας έχει νόημα, σε άλλες δεν έχει και θα πρέπει να υπάρξει ευελιξία. Κάτι άλλο που τέθηκε, το κόστος των προτάσεων έργων. Και προς τα εκεί στρέψατε την προσοχή σας όταν μας ρωτήσετε ότι μήπως όλες αυτές οι απαιτήσει αποτρέπουν και αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις. θυμάμαι ότι από τη Βρετανία είχα τεθεί συχνά τα ερωτήματα από επιχειρήσεις που λέγανε έχει νόημα να ζητήσουμε, να το κάνουμε μόνοι μας ή μήπως είναι καλύτερα να ζητήσουμε από ένα consulting να μας τι κάνει την πρόταση γιατί αυτή παρά είναι περίπλοκη για μας. Και εν τέλει το ερώτημα είναι αξίζει όλη αυτή η διαδικασία για να πάρουμε μια επένδυση. Εκεί υπάρχουν επιφυλάξεις. Η εμπειρία μας πάντως λέει ότι οι αμφιβολίες αυτές περιορίζονται σε περιοχές που έχουν την πολυτέλεια να αντλήσουν πόρους από άλλες πηγές ή όταν είναι υγιείς επιχειρήσεις και μπορούν να αντλήσουν πόρους μόν, μόνος τους. Εμείς βρισκόμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει αυτό το λουξ. Στην κεντρική Ισπανία παρακολουθούν με θρησκευτική ευλάβεια το τι γίνεται στα διαφθορτικά ταμεία. Τώρα, ποιος πρέπει να προωθήσει τη βιωσιμότητα. Κοινή προσπάθεια πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρχουν και σωστές οδηγίες από, την το ευρωπαϊκό επίπεδο. Προφανώς όμως, η ο επισπεύδων, η πρωτοπορία πρέπει να προέρχεται από το κράτος μέλος. Εκεί είναι που υπάρχουν οι προτάσεις και υλοποιούνται τα πράγματα. Ο ρόλος του ελεκτικού συνεδρίου. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν είναι κάποιος εδώ από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Εμεί είδαμε πολύ προσεκτικά την το εγχειρίδιό τους για τον έλεγχο επιδόσεων. Δεν υπάρχουν πολλά για τη βιωσιμότητα, παρότι είναι πολύ καλό κείμενο. Τονίζει τον αντίκτυπο την αποτελεσματικότητα, δεν τονίζει την διάρκεια. Νομική βάση. υπάρχει μία τάση να κάνουν τα κράτη-μέλη την νομοθεσία επιχρυσωμένη, δηλαδή κάπως να την, ε, να, προσπαθούν να τη βελτιώσουν. Εμείς δεν ρωτήσαμε τις διαχειριστικές αρχές, τι επιπτώσεις έχει το αυτό σε εθνικό ή ε, σε περιφερειακό επίπεδο. Best practice examples you mentioned. Παραδείγματα βέλτιστης της πρακτικής. Εμείς έχουμε στη μελέτη κάποια παραδείγματα επιχειρήσεων. Προσπαθούμε να δείξουμε και να τις ρωτήσουμε δηλαδή για να το δείξουμε τι διαφορετικό έκαναν, πώς επιβίωσαν μετά την πενταετία. Και η βάση δεδομένων, αν τη δείτε, σε όλες τις γενικές ευθύνσεις υπάρχουν βάσεις δεδομένων βέλτιστων πρακτικών. Και αν τις δείτε από πλευράς επιχειρήσεων, ε, θα διαπιστώσετε ότι είναι επιφανειακές. Δηλαδή δεν σου λένε, σου δίνουν ωραία παραδείγματα, αλλά δεν σου λένε τι πρέπει να κάνει στην ουσία. Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές πρέπει να ενισχυθούν πιστεύω περισσότερο με πολύ συγκεκριμένη περιγραφή σε σχέση με το κριτήριο βιωσιμότητας. Τι εμπειρίες υπάρχουν, τι μπορεί να γίνει για να το πετύχουμε. Υπάρχουν εμπειρίες που μπορούν να μεταφερθούν. Νομίζω ότι η μελέτη βέλτισης πρακτικής που έχουμε είναι περιορισμένες, μία σελίδα το πολύ. Τώρα πρέπει να μεγαλώσουν πιστεύω. Για την... Δεν κατάλαβα την ερώτησή σας για το θέμα της επιβολής προϋποθέσεων, του conditionality, όπω λέμε. Δεν ασχοληθήκαμε πάντως με το θέμα αυτό στην ε, μελέτη. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Αγγελάντ, τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι επικεφαλής της ε, ομάδας λειτουργικής, ε, επιχειρησιακής μάλλον ε, αποτελεσματικότητας υπεύθυνο και για την εφαρμογή του άρθρου 57 μεταξύ άλλων. Από την Κομισιόν πρέπει να πω ότι καλωσορίζουμε αυτήν την μελέτη και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή βοήθεια για την διάρκεια και την αποτελεσματικότητα των projects ε, και ε, βεβαίως ε, θεωρούμε ότι και το πλαίσιο, τα συμπεράσματα λέει, τα οποία προκύπτουν από την μελέτη αυτή συμπίπτουν και με το επόμενο πολιετές πλαίσιο. Από την πλευρά της Κομισιόν καλωσορίζουμε και τις παρατηρήσεις όσον αφορά την βοήθεια προς μεγάλες εταιρείες παρατηρήσεις ε, οι οποίες ε, εν πολλής ευθυγραμμίζονται και με, τις, ε, με την επιχειρηματολογία που έχει αναπτύξει η Κομισιόν εξ αρχής. ενδεχομένως πηγαίνουν προς μια λίγο διαφορετική κατεύθυνση οι εξελίξεις ε, του νομοθετικού πλαισίου, αλλά πάντως θεωρούμε ότι αυτά που αναφέρονται στην μελέτη ε, ε, επιβεβαιώνουν τα συμπράγματα της Επιτροπής για τις μεγάλες εταιρείες. Είναι γεγονός ότι ένας μεγάλος βαθμός της αιστείας σχετικά με το άρθρο 57 μέχρι τώρα έγινε στην ε, διασύνδεση με την εντοπιότητα ε, και e funding. Um, particularly easy to stop delocalization. Ε, ε, και η μετακίνηση, το πρόβλημα αυτής της μετακίνησης της παραγωγής ε, που μπορεί να γίνει και μέσω χρηματοδότησης με ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουμε κάποια συγκεκριμένα, κάποιες συγκεκριμένες επιπτώσεις όπου επιτυχώς αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα αυτό σε σε τούτη την προγραμματική περίοδο και ελπίζουμε ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο μηχανισμό, καλύτερο μηχανισμό έτσι ώστε να γίνει ακόμα πιο δύσκολο να γίνει αυτή η μετατόπιση. Υπάρχουν και κάποια άλλα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί όσον αφορά την ε, περιπλοκότητα ε, της ε, μεγαλύτερης ε, αηφορίας και πιο γρήγορα. Νομίζω ότι αυτό είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Έχουμε τη διαδικασία της την διαδικασία την αρχική της πρόσκλησης ενδιαφέροντος που πρέπει να είναι αρκετά ελκυστική έτσι ώστε να δημιουργήσει ενδιαφέρον αλλά από την άλλη πλευρά ε, έχουμε, πρέπει να έχουμε και την επόμενη φάση έτσι ώστε να μπορεί να γίνει μια σωστή επιλογή ανάμεσα από όλα τα ε, προγράμματα τα οποία θα έχουν υποβληθεί. Ε, και επομένως ναι θα πρέπει να υπάρξει μια περαιτέρω εξισορρόπηση αλλά νομίζω ότι στα κράτη των κρατών μελών και μάλιστα των περιφερειών ε, των κρατών μελών εκεί βρίσκεται, στο χέρι τους βρίσκεται το μπαλάκι. Εμείς θέλουμε να υπάρξει απλούστευση έτσι ώστε να μην έχουν κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεγάλο βάρος ε, και αυτό θα υπογραμμίσουμε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που ξεκινούν ε, τώρα και βεβαίως και στη διάρκεια των ε, επιτροπών επιθεώρησης monitoring committees που θα ακολουθήσουν. Πρέπει να σας πω και δεν θα εκπλαγείτε ε, ότι χαιρόμαστε γιατί ε, υπάρχει αυτή η νομική σαφήνεια την οποία έχουν αναγνωρίσει ε, και τα κατατόπους ελεγκτικά συνέδρια ε, πάντως ε, οι ε, διαχειριστικές αρχές θεώρησαν ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλη διαφάνεια ή σαφήνεια κατά την άποψη των κατατόπους διαχειριστικών επιτροπών. Εγώ νομίζω ότι οι διαχειριστικές αυτές επιτροπές θα πρέπει να ε, προσπαθήσουν να ε, κάνουν στους δικαιούχους πιο κατανοητά κάποια στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να προχωρήσει ο ε, κανονισμός έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς από τη δική μας πλευρά μεγάλη σημασία δίνουμε στο να εξηγήσουμε σαφώς το τι πρέπει να κάνουν και στην ε, ε, ε, διάρκεια της υποβολής υποψηφιότητας και αργότερα το τι πρέπει να κάνουν δηλαδή αυτές οι επιτόπου διαχειριστικές αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για να κλείσει ο Μάρκους Πίπερ έχει το λόγο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό που κατέστησα φες και από τη μελέτη και από τις συζητήσεις είναι η σπουδαιότητα του θέματος. Θα ήθελα το Κοινοβούλιο να λαμβάνει υπόψη του σοβαρότερα τις διαπιστώσεις αυτές. Όταν έχουμε μπροστά μας μεγάλες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε να παίρνουν πόρους διότι είναι σαν, σαν ηλεκτρική σκούπα, ρουφάνε τους πόρους. Ενώ η απόδοση είναι λιγότερο ε, θετική, λιγότερο αποτελεσματική από ό,τι σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Τώρα το θέμα της μετακίνησης επιχειρήσεων. Η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει κάπως ε, μεγαλύτερη επίγνωση του προβλήματος. Δεν μπορεί μετά από πέντε χρόνια να σταματάει ας πούμε η λειτουργία των πόρων. Οι επιχειρήσεις που μετακινούνται δεν θα πρέπει να μπορούν να ε, παίρνουν κονδύλια από τα διαδοτικά ταμεία. Το έχουν πει κάποιοι ευρωβουλευτές αυτό. Είμαι βέβαιος ότι δεν έχουμε καταλάβει απόλυτα το μέγεθος του προβλήματος έχουμε, καταλαβαίνουμε το φαινόμενο αυτό όταν υπάρχει ένα ανώτατο όριο, αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν φύγει εκατοντάδες επιχειρήσεις αφού, ε, μετά, αφού πήραν ενισχύσεις. Πάντως ε, η μελέτη ήταν χρήσιμη την κυρία Χολμάγερ, δεν νομίζω όμως ότι είναι επαρκής για να ε, βεβαιωθεί ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ενισχύσεις των διαδοτικών ταμείων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ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 αν κανονικά δεν υπήρχε πρόβλημα, ήταν εδώ ο κύριος Τσβίκη από το Ελεκτικό Συνέδριο. Δεν ξέρω αν είναι εδώ ο κύριος Τσβίκη. Το ψάχνουμε. Ε, Υπάρχει ο εκπρόσωπος του Ελεκτικού Συνεδρίου. για να πάμε σε αυτό το σημείο της μέσης διάταξης πρέπει να έχουμε παρόντα τον εκπρόσωπο του ελεκτικού συνεδρίου που ασχολείται με το θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ημερησία διάταξη. Τι θέλετε κύριε Μαρινέσκου. Αν κατάλαβα καλά έπρεπε να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη γιατί η κυρία Γιάλα Σέντερ δεν ήταν στην αίθουσα αλλά μια και είναι εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ δεν ζήτησα πραγματικά να αλλάξει η μεσαία. Είπα ότι είμαι διαθέσιμο, εάν έλειπε η κυρία Γιάννα Σέντερ. Ναι, να περιμένουμε να έρθει εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου και να μιλήσει η κυρία Γιάννα Σέντερ. Okay. Uh... A να fogalmaztam, akkor az én Συγγνώμη, το είπα γιατί το νόμιζα ότι ο κύριος Μαρινέσκου το είχε ζητήσει, αφού δεν... Ε, υπάρχει ζήτημα αλλαγή τη ημερήσια διάταξη γιατί ήρθε η κυρία Γιάλα Σέντερ. Δεν αλλάζουμε λοιπόν τη ημερήσια διάταξη και προχωράμε στο σημείο 11. τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα τη της επιβολής του νόμου, δηλαδή τη Europol. αποφασει 2009 2009-371 GHA και 2005-681 GHA. Η κυρία Γιάλα Σέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και τον κύριο Μαρινέσκου για την δυνατότητα για την, ε, τέλος πάντων, ε, γιατί έδειξε ότι ήταν ευέλικτος. Ξέρετε, τέτοια εποχή που είναι, δεν ξέρουμε τι αυτά είναι το αεροπλάνο. Τέλος πάντων, εγώ είμαι εδώ. Έχουμε την υποχρέωση να δώσουμε γνωμοδότηση της Επιτροπής μας προς την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών για την Europol, τον κανονισμό που παρουσιάζει η Επιτροπή για να ενημερώσει και να προσαρμόσει στις νέες απαιτήσεις την Europol. Ο οργανισμός αυτός, είχαμε πληροφορίες άλλωστε πολύ σημαντικές και ε, τους τελευταίους μήνες και τις τελευταίες εβδομάδες στην, Ελλάδα, στην Ισπανία αλλά και αλλού για την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα της Ευρωπόλ που έχουν ε, εντολή από τη συνθήκη να ενισχύσει όχι μόνο την αστυνομική συνεργασία αλλά να το κάνει και εν ώψη μιας προοπτικής διαμόρφωσης στην Ένωση ποινικού δικαίου. Είδαμε πρόσφατα τη συζήτηση για όλο αυτό το ποινικό και πλαίσιο, το ποινικό μέλλον της Ένωσης. Η γνωμοδότηση που σας παρουσιάζω προσπαθεί με μια σειρά τροπολογιών να ενισχύσει το ρόλο του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας στην παρακολούθηση της εφαρμογής, της αποτελεσματικής εφαρμογής του προπολογισμού του οργανισμού στην εκπλήρωση των καθηκόντων του. Θα γνωρίζετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συζήτηση στα πλαίσια της απαλλαγής της φετινής χρονιάς έκθεση μπράντι διότι η Επίτροπη μας ε, πρότεινε, σύστησε, με μια γενική σύσταση λόγω της οικονομικής, ε, των οικονομικών περιστολών, μείωση των δαπανών για τη Europol και την C-Pol επειδή είναι και αστυνομία θα καλεί ο καθένα, είναι και κοντά μεταξύ τους, ήταν σκόπιμο να συγχωνευτούν. Εγώ μίλησα με την κυρία Γκερμπράντη, με τον κύριο Γκερμπράντη και μου εξήγησε το ενδεχόμενο να μετακινηθεί και η ΣΥΠΟΛ στην Χάγη. Η ιδέα ήταν όπως και για άλλους οργανισμούς να μην ξεκινήσουμε κομμάτι-κομμάτι αλλά να το κάνουμε όλα μαζί. Η ομάδα μου την εποχή εκείνη είχε εκφραστεί αντίθετα ε, με την συγχώνευση δύο οργανισμών που είχαν διαφορετικά καθήκοντα, που δημιουργήθηκαν διαφορετικούς σκοπούς και που επειδή ακριβώ πρόκειται για αστυνομική δράση και μάλιστα ευρωπαϊκή αστυνομική δράση, θεωρήθηκε ότι είναι ένα λεπτό ευαίσθητο ζήτημα και έπρεπε να εξετασθεί πιο προσεκτικά. Η άποψή μας είναι αυτή που ήταν και την εποχή της απαλλαγής. Οι δύο οργανισμοί έχουν διαφορετικές εντολές, παρότι η πελατεία τους είναι παρόμοια. Δεν είναι η ίδια. Πάντως τα καθήκοντα και οι ευθύνε τους είναι διαφορετικές. Η ιδέα λοιπόν να διαμορφωθεί, να συγχωνευτεί η Europol που έχει και νέες ευθύνε με έναν οργανισμό όπως η ΣΥΠΟΛ που έχει περίπλοκη εντολή και πως στόχος της είναι η κατάρτιση, είναι σε άλλη γραμμή του προπολογισμού για παράδειγμα, θεωρήθηκε κάπως πρόημο η πιθανή εξοικονόμηση που θα μπορούσε να προκύψει όταν συζητήσαμε την Επιτροπή με τους υπεύθυνου, με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών και από την Επιτροπή Προϋπολογισμών με οδήγησε στο συμπέρασμα και φαίνεται στις τοπολογίες ότι δεν καταλαβαίνω κατά πόσον η συγχώνευση των δύο υπηρεσιών θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερα, περισσότερα πλεονεκτήματα από ό,τι προβλήματα. Διότι η Europol σε αυτή τη νέα εντολή που έχει χρειάζεται να σταθεί στην ανάπτυξη των βασικών της καθηκόντων. Όπως το λέει και η συνθήκη. Ενώ η ΣΥΠΟΛ ασχολείται με την κατάρτιση. το Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση της Βρετανίας μας λέει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ε, υπηρεσία που βρίσκεται στην, στην Βρετανική Αστυνομική Ακαδημία. Η Επιτροπή, όπως και με άλλους οργανισμούς, όταν ολοκληρώνεται η σύμβαση, ε, όταν ολοκληρωθεί η σύμβαση δηλαδή η ενική, θα λάβει τις, αποστάσεις, τις αποφάσεις της και θα δούμε τότε τι θα γίνει. Ο κανονισμός τώρα της Europol είναι κάτι που πρέπει να μας αποσχολήσει ξέχωρα. Τώρα, βάσει και της εντολής επιτροπή στην απαλλαγή, υπέβαλε την τροπολογία υπαριθμών 8. σε συνεργασία με την Επιτροπή που μου είπε ότι αρχικά δεν σκεφτόταν τη συγχώνευση. Η ιδέα επιβλήθηκε το Ποντινά ή επιταχύνθηκε από την ανάγκη περικοπών που δεν είναι πάντα καλή σύμβουλος όταν μιλάμε για θέματα όπως την αστυνομική συνεργασία στην Ευρώπη. Όταν προσπαθούμε να υλοποιήσουμε το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο haya sinergias entre las agencias, ahí donde pueda haberlas, entre las dos agencias. Λοιπόν, η συνεργασία των αστυνομικών αρχών είναι σημαντική και εκεί τονίζουμε ότι τα κοινωνίζουν τα πιο σημαντικά σημεία. Κατόπιν παρουσίασα μια σειρά τροπολογιών όπου όπως προκύπτει και από την πρόταση επιτροπής και από την ανάγκη συγχώνευσης, εμφανίζεται μια εκτελεστική επιτροπή που προτείνει επιτροπή, τις οποίες τα καθήκοντα είναι ακριβώς τα ίδια με του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που τα διαχωρίζει. Εγώ δεν βλέπω την ανάγκη για κάτι τέτοιο. Ας μας το εξηγήσει καλύτερα η Κομισιόν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω γιατί πρέπει να υπάρχουν δύο όργανα που είναι στην ουσία ταυτίζονται. Η απεκάλυψη δραστηριοτήτων θα μπορούσε να δυσκολέψει τη διαχείριση. Επίσης εμφανίζεται και η σχέση μεταξύ Europol, Just και Όλαφ. Εγώ διατήρησα την... το σχετισμό που επιβάλλει και η συνθήκη για τις σχέσεις Europol, Eurojust που υπάρχει όπου έχουν μια σχέση αμοιβαιότητας. Η... η υλοποίηση τη αστυνομική συνεργασίες που επιβάλλει η συνθήκη και τα θέματα ε, ανταλλαγής δεδομένων να απαιτεί τη συνεργασία με το Eurojust και το αντίστροφο, να μπορεί δηλαδή η Eurojust να δουλέψει με τα στοιχεία της Europol. Για την Όλαφ, φαίνονται και στις τροπολογίες, θέλουμε να διαφυλάξουμε το βασικό στόχο της Όλαφ σε σχέση με τον οργανισμό, δηλαδή την καταπολέμηση της απάτης ή των λανθών που εφαρμόζονται σε, στην υλοποίηση διοικητικών κανονισμών. Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να μετατρέψουμε τα καθήκοντα της Όλαφ σε καθήκοντα Ευρωπαϊκής Αστυνομίας. Έχει ξεχωριστεί αρμοδιότητα η Όλαφ που σχετίζονται με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ενώ το Eurojust και η Europol έχουν στόχο όπως σας είπα την ενίσχυση και υποστήριξη του μελλοντικού ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου. Κάποιες άλλες τροπολογίες έχουν στόχο να ενισχύσουν τα καθήκοντα του εκτελεστικού, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, την, το, το θέμα της σύγκρουση συμφερόντων. Στη διαχείριση αυτή, ο εκτελεστικός διευθυντής της Europol, στο, μάλλον σε ό,τι αφορά τον εκτελεστικό διευθυντή της Europol, ζητώ να υπάρχει παρακολούθηση της δράσης του και από το Κοινοβούλιο. Αυτά είναι όλα. Περιμένω τις απόψεις σας και βεβαίως παραμένω ανοιχτή σε κάθε ενδιαφέρουσα και θετική ιδέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ingeborg. Ευχαριστώ πολύ. Τι να σας πω. Αυτό πλέον έχει γίνει σύριαλ. Εδώ και χρόνια ζητούμε την ε, ε, ένωση ας πούμε της Europol με την ε, Σέπολ. Κυρίως γιατί η Σεπόλ είναι μικρή οργάνωση. Ίσως είναι η πιο μικρή, ο πιο μικρός οργανισμός που έχουμε. Αλλά παρότι είναι μικρός οργανισμός θα πρέπει να έχει ένα ολόκληρο διοικητικό δυναμικό όπως ε, οφείλει κάθε οργανισμός. Γι' αυτό ζητήσαμε τη συγχώνευση. Έτσι ώστε η διοίκηση να είναι κοινή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, η ΣΕΠΟΛ να είναι χωριστός οργανισμός, έστω και αν ο διευθυντής της ε, βεβαίως για τους δικούς του λόγους επιθυμεί να παραμείνει χωριστός οργανισμός ε, και μάλιστα ε, και επειδή και το προσωπικό προτιμά να μείνει στο Λονδίνο και όχι να φύγει από το Λονδίνο και να πάει στις κάτω χώρες. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να εγγραφεί στο ευρύτερο πεδίο, στην ε, ευρύτερη χωροταξία κατά κάποιο τρόπο των οργανισμών. Γιατί σήμερα το πρωί λέγαμε που θα καταλήξουμε αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Γιατί θα φτάσουμε σύντομα στα όρια της κατηγορίας 5. Πόσο σοβαροί μπορεί να είμαστε ε, στην ε, βούληση αλλαγής. Νομίζω ότι εδώ ε, παίζεται κατά κάποιο τρόπο η θέληση, η βούληση να κάνουμε αλλαγές και η ικανότητα δράσης που έχουμε. Ε, τα, κράτη-μέλη από τη μία μεριά μαλλιοτραβιούνται ε, για τις ε, δομές των Βρυξελών και από την άλλη πλευρά στυλώνουν τα πόδια τους και δεν θέλουν καμία αλλαγή όσον αφορά τις υφιστάμενες δομές. Θα είναι πολύ μεγάλο λάθος εάν και εφόσον το Κοινοβούλιο υποστηρίξει τα κράτη-μέλη σε αυτήν τους ε, την ε, κίνηση. Θα πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη τάση συγχώνευσης ε, των οργανισμών. Europol, Sepol λοιπόν, είναι πολλοί αυτοί που είναι υπέρ της συγχώνευσης και πολλοί που είναι κατά. Ας προσπαθήσουμε να δούμε λίγο από απόσταση τα πράγματα, θα διαπιστώσουμε ότι λόγω προβλημάτων διοικητικής διαχείρισης ένας μικρός οργανισμός στην ουσία ο ίδιος θα έπρεπε ε, να ζητήσει την βοήθεια ενός μεγαλύτερου οργανισμού. Στο Λονδίνο ξέρουμε ότι η σύμβαση λύγει σε λίγο. Τι θα κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση. Θα αρχίσουμε να ψάχνουμε για νέα μίσθωση γύρω από το Λονδίνο ξέροντας ότι είναι πάρα πολύ ακριβά και τα ενίκια και όλα ή θα ε, ε, ε, ζητήσουμε να υπάρξει συγχώνευση. Εδώ και χρόνια έχουμε εκφράσει την επιθυμία για τέτοια συγχώνευση αλλά βεβαίως θα πρέπει να δείξουμε και ένα ελάχιστο θάρρος. Ήμουν ε, παρούσα ε, σε μια προηγούμενη ε, συνεδρίαση για τη συγχώνευση των οργανισμών και η Ιούτα Χάιγκ της σοσιαλιστικής ομάδας, της ομάδας των σοσιαλιστών και δημοκρατών ήταν υπέρ της συγχώνευσης. Δεν ισχύει λοιπόν αυτό που μας είπες. Δεν ισχύει ότι όλοι είχαν την ίδια άποψη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, εάν η κυβέρνησή μου κάνει λάθος, ε, να αντιταχθώ σε αυτήν τη λάθος ε, θέση της κυβέρνησης. Νομίζω, ε, ε μας λένε, μπορούμε να συνεργαστούμε περισσότερο, αλλά δεν μπορούμε να συγχωνευτούμε ή δεν θέλουμε να συγχωνευτούμε. Εάν δεν μπορούμε να πούμε σε έναν διευθυντή ε, ότι καλά προσπάθησε και θα δούμε τι θα γίνει, δεν είναι σωστή αντιμετώπιση. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε να περνάνε ε, τέτοια χονδροειδή πράγματα και να μην ε, αντιδρούμε θα πρέπει να παρακολουθήσουμε από κοντά ε, το θέμα. Εγώ συμφωνώ και στηρίζω απολύτως την πρόταση της ε, Κομισιόν γιατί στην ουσία ταυτίζεται με αυτό που ε, πολλά χρόνια απαιτεί και ζητά η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή με τη στήριξη των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Νομίζω ότι εδώ παίζεται ό,τι μας έχει απομείνει από την αξιοπιστία μας και θα πρέπει η πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή μας ελέγχου του προϋπολογισμού. Weil wenn wir das auch nicht wollen, dann kann ich nur sagen, werdet ihr staunen, werdet ihr staunen, welche Kosten να προσπαθήσουμε λοιπόν να ξαναδούμε τη συνολική χωροταξία των οργανισμών γιατί διαφορετικά θα έχουμε τον, ε, στο επόμενο χρονικό διάστημα έκρηξη των δαπανών, ε, του κόστους λειτουργίας των οργανισμών αυτών. Εγώ στηρίζω λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και δεν μπορώ να στηρίξω τις προτάσεις τροποποίησης της εισηγητρίας. Καλό δε όλους τους συναδέλφους να σκεφτούν πολύ σοβαρά. τα διακυβεύματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και πολύ σοβαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από τη στιγμή που γίνεται λόγος ε, για ε, συγχώνευση, οποτεδήποτε μιλάμε για συγχωνεύσεις, τα πράγματα είναι οδυνηρά. Όμως Πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος δεν έχει πολύ μεγάλη ε, επίπτωση όσον αφορά τον προϋπολογισμό. E, e, είναι γεγονό ότι έχουν ξεκινήσει καταστάσεις 20 χρόνια πριν. Ε, ε, Βεβαίως, ε, ίσως πρέπει να ξαναδούμε λίγο τη χωροταξία αυτών των οργανισμών, αλλά θα πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν. Και βεβαίως ε, προκύπτει και το μέγα ερώτημα για το Στρασβούργο. Γιατί γίνεται λόγος εδώ για το κόστος, αλλά το κόστος για το οποίο συζητάμε εδώ είναι, ξέρω εγώ, 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για τα λίγα και να μην μιλάμε για τα πολλά. Ε, θα πρέπει να μετρήσουμε, να ζυγίσουμε τα πράγματα, να δούμε ποια είναι τα πολιτικά ζητήματα, ε, να δούμε ποια είναι η πραγματική επίπτωση της κάθε απόφασης στον ε, προϋπολογισμό. Βεβαίως ε, μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικός ο τρόπος λειτουργίας αυτών των οργανισμών και να δουλεύει. Να λειτουργούν μεταξύ τους με καλύτερη ε, συνεργασία. Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Charles Williams. Έχετε το λόγο. Κομισιόν παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν ε, αναφερθώ στο ζήτημα της συγχώνευσης ήμι, να περάσω στο θέμα του εκτελεστικού συμβουλίου που ανέφερε ο εισηγητής. Η εισηγητρία. Το εκτελεστικό συμβούλιο είναι πράγματι ένα όργανο το οποίο θα δρά μεταξύ των ε, τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό ακολουθεί την κοινή προσέγγιση και τις ε, σχετικές ε, κατευθύνσεις που δίνονται εκεί πέρα. Επίσης πρέπει να πω πως η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει πως υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ενός τέτοιου εκτελεστικού συμβουλίου, δεν είναι απαραίτητο. Και τέλος να πω πως η Κομισιόν έχει σημειώσει τα όσα είπε ο εισηγητής ε, για την πρόταση αυτή. Να έρθουμε τώρα στο ζήτημα των ε, συγχωνεύσεων. Η Κομισιόν παρουσίασε μια πρόταση να συγχωνευτούν οι δύο αυτές αποκεντρωμένες υπηρεσίες είναι ακόμα επιτάπητος αυτή η υπηρεσία. Η Κομισιόν δεν έχει κάνει άλλη πρόταση μέχρι στιγμή και να σας πενθυμίσω γιατί έγινε αυτή η πρόταση. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε πως μπορεί να υπάρξει κάποια συνέργεια με το να συγχωνευθούν όλα τα της δημοσίας τάξεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια υπηρεσία από την στήριξη μέχρι την ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών, μέχρι την, τον υποστηρικτικό ρόλο της εκπαίδευσης της ΣΕΠΟΛ. Γι' αυτό θεωρούμε πως πρέπει η ΣΕΠΟΛ να γίνει μια Ακαδημία της Ευρωπόλ. Θεωρούμε πως ε, έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε και πιο ουσιαστική εκπαίδευση και πιο επιχειρησιακή. Κατόπιν υπάρχει το ζήτημα του κόστους. Θεωρούμε πως μέσω του να μην υπάρχει διπλή διοικητική υποστήριξη θα κάνουμε κάποια οικονομία οικονομία η οποία θα έχετε δει στην ε, πρόταση ε, η οποία θα σημαίνει πως τα κονδύλια αυτά θα ξαναπάνε προς ε, τους ε, σκοπούς της εκπαίδευσης. Αυτή ήταν μια ανακοίνωση που εκδώσαμε μαζί με την νομοθετική πρόταση και είναι κάπως πιο δομημένη για το πώς μπορεί η Κομισιόν να δει καλύτερα τις πτυχές της εκπαίδευσης. Θεωρώ πως για να εφαρμόσουμε πλήρως τις φιλοδοξίες μας θα χρειαστούμε το ισοδύναμο 12 θέσεων προσωπικού πλήρους απασχόλησης και αυτό σημαίνει βεβαίως πως θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη μείωση προσωπικού άλλη και αυτό μπορεί να γίνει με τον τρόπο που περιέγραψα. Οπότε δεν γίνονται οικονομίες για το τίποτα, αλλά θα βοηθήσουν την βελτίωση της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων στον τομέα της ε, επιβολής του νόμου. Τέλος, ε, Πέρσι υπήρχε και η κοινή προσέγγιση των τριών θεσμικών οργάνων που ευθύθηκε για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και βεβαίως η Κομισιόν την κατέστησε πιο επιχειρησιακή τον Δεκέμβριο και τώρα έχουμε την πρώτη νομοθετική πρόταση που στόχο έχει να λάβει υπόψη πλήρω αυτές τις σκέψεις. Που είχαν βεβαίως στηριχθεί ε, ευρύτατα στο διοργανικό αυτό έγγραφο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και την Επιτροπή για τα σχόλια. Να υπενθυμίσω ότι στο θέμα των υπηρεσιών ευτυχώς το, μάλλον, το κοινοβούλιο λειτουργεί σαν γιογιό. Με το που κάτι θέλει να βγάλει από τις αρμοδιότητες επιτροπή, τσαφ, πετάμε μια υπηρεσία, αλλά μετά μετανιώνουμε και αποφασίζουμε το ξαναβάλουμε στην κοινότητα. Δηλαδή μπαίνουν οι αρμοδιότητες, βγαίνουν από την επιτροπή. Αυτό είναι αρνητικό και για τους πολίτες και για την καλή διαχείριση από πλευράς του Κοινοβουλίου. Δεν νομίζω ότι ο τρόπο λειτουργία είναι σωστό, Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά και με σαφή τρόπο τα καθήκοντα κάθε οργανισμού. Μεταξύ αυτών μιλάμε και για τις δομέ των Βρυξελών. Δυστυχώ, δεν μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για τις Βρυξέλλες και τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ε, παρουσιάζουν, δυστυχώς ή ευτυχώς, την ε, δραστηριότητα της Ένωσης επιτόπου. Έκλεισε, αποφάσισε ο κύριος Κάμερον, η κυβέρνηση του κύριου Κάμερον να κλείσει την, ε, να μην πάνω ότι δεν ενδιαφέρεται για την ΣΥΠΟΛ και αυτό είναι δείγμα και της αύξησης του αντιευρωπαϊσμού στη χώρα αυτή. Αυτό δεν συμβαίνει αλλού. Όταν σκεφτόμαστε λοιπόν τι καθήκοντα, τι εντολή και τι αποτελεσματικότητα και ικανότητα θα έχουν οι υπηρεσίε αυτές, θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι δεν είναι η εποχή περικοπών. Δεν θα ήταν σοβαρό βέβαια να νομίζουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση και ενόψη των εκλογών να κόβουμε, να περικόπτουμε μία υπηρεσία μόνο και μόνο γιατί η λέξη «πολ» είναι και στις δύο υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες υπάρχουν στις κράτη-μέλη για να δείχνουν την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι αυτές οι υπηρεσίες, αυτές οι δομές έχουν δημιουργήσει πολύ, καλή, πολύ καλό δίκτυο μεταξύ τους που δεν ε, έχει ούτε κάνει η Επιτροπή. Δηλαδή έχουν δημιουργήσει μια επικοινωνία μεταξύ τους πολύ καλή που μπορούν να βελτιώ, επιτρέψουν τη βελτίωση ε, του συντονισμού χωρίς να κλείσουμε τα, ε, τις δομές αυτές. Σε μια περίοδο εκλογών δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να το να το περάσουμε. Γιατί η Europol. Η εντολή που έχει η Europol είναι εξαιρετικά λεπτή. Είναι η εντολή που της δώσαμε να ανοίξει το κέντρο της μάχης κατά της εγκληματικότητας, μία από τις μεγάλες προκλήσεις της Ένωσης. Εγώ θα προτιμούσα λοιπόν να ασχοληθεί η Europol με αυτό που της είπαμε να κάνει. Και τι της είπαμε να κάνει. Αυτά που λέει και η συνθήκη. Θα ζητούσα λοιπόν από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής να μου πει το εξή. Η συνθήκη αυτή καθεαυτή παρέχει την επαρκή νομική βάση για να ασχοληθεί η Europol και με την ε, παροχή μαθημάτων κατάρτισης. Εγώ έχω επιφυλάξεις. Δεν ξέρω αν αυτές τις επιφυλάξεις τις έλυσε η Επιτροπή. Επίσης, η Επιτροπή στην εξήγηση της πρότασής της λέει ότι η συγχώνευση, η πλήρη συγχώνευση σε Πολ και Europol δημιουργεί συνέργεια, γλιτώνει κάποια χρήματα για την περίοδο 15-20, αλλά στην επόμενη παράγραφο λέει παρότι η Europol χρειάζεται, θα χρειαστεί περαιτέρω πόρους για να υλοποιήσει τα νέα καθήκοντα που σχετίζονται με την κατάρτιση των αστυνομικών υπαλλήλων και διάφορα άλλα. Δηλαδή, έχει η Επιτροπή και μας λέει θα κόψουμε κάτι θα περιορίσουμε κάτι, αλλά λέει τι επιπλέον δαπάνες θα υπάρχουν. Αν τελικά η προσταφαίρεση βγάζει μηδέν και ο μόνος στόχος είναι να έχουμε μία, έναν οργανισμό λιγότερο και άκουσα κάποιους να λένε ότι είναι online η κατάρτιση. Όχι, δεν είναι. Η κατάρτιση αυτή γίνεται σε τόπους όπου η αστυνομία δουλεύει ήδη. Και η της πόλη είναι από τις ε, ε, καλύτερες ε, δομές κατάδυσης. Εγώ στην Κρίν είχα δει πως δουλεύει η γεωδοπολή, είχα μείνει αποσβολωμένη. Εγώ λοιπόν δεν θα έλεγα τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε να λόγω περικοπών να, να αλλάξουμε τις εντολές οργανισμών που δεν είναι στι Βρυξέλλε, που είναι σε κράτη-μέλη. Είναι, δηλαδή που είναι αυτό που βλέπουν οι πολίτες από την και που λειτουργήσαν καλά. Είχε προβλήματα η ΣΕΠΟΛ, αλλά δεν νομίζω ότι είχε ε, προβλήματα υπαρξιακά. Τα προβλήματα διορθώθηκαν. Άλλη εντολή έχει η ΣΥΠΟΛ, άλλη έχει η Europol. Δεν έχει να κάνει η Europol με την κατάρτιση αστυνομία. Η πρόκληση Άλλο είναι ο στόχος της, να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα. Όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Η κυρία Χάουγκ, συνάδελφος, μην δουκαριζόμαστε, ε, την ίδια, την ίδια εθνικότητα έχετε και εσείς κύριε Γκρέσλερ, στις 22 τονίζει, στις 22, θα τονίσει μάλλον στις 22 Σεπτεμβρίου την άποψή της, δικό της θέμα είναι, ε, υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που δεν έχουν την ίδια άποψη με την κυρία Χάουγκ. Εγώ θα προτιμούσα λοιπόν να μην τρέχουμε να αλλάζουμε τώρα τα καθήκοντα των υπηρεσιών που συνεχίζουν να είναι ένα στοιχείο που παρουσιάζει την Ευρώπη στους πολίτες και θα ζητούσα από την Επιτροπή Πρόεδρε να μας διευκρινίσει κατά πόσο η συνθήκη δίνει την επαρκή νομική βάση στην ε, Europol για τα νέα καθήκοντα που θέλει να τη δώσει η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Nem vettem észre előbb Greszle képviselő asszony jelentkezést. Δεν βλέπω να... Α, παρατήρησα πως ε, τον λόγο ζήτησε και η κυρία Γκρέσλε. Πριν ξέρω στο λόγο, θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία στον εκπρόσωπο της Κομισιόν ε, αν θέλει να αντιδράσει σε αυτό το είπε η κυρία Γιάλα Σέντερ. για το συγκεκριμένο ερώτημα για τη νομική βάση. Πράγματι, το άρθρο 89 ε, της συνθήκης πράγματι είναι αυτό το οποίο καθορίζει τα της Ευρωπόλ. Εκεί πέρα υπάρχει, παραδείγματος, υπάρχουν διάφορες ιδιαιτερότητες όπως ο κοινοβουλευτικός έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια η αρμοδιότητα για εκπαίδευση είναι κάτι το συμπληρωματικό, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα για την εκπαίδευση του προσωπικού. Η άποψή μας είναι πως δεν υπάρχει κάτι στη συνθήκη το οποίο απαγορεύει στην Ευρωπόλ ε, σύμφωνα με το άρθρο 88 εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και τα μέσα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την εκπαίδευση του προσωπικού αλλά βεβαίως ε, ομολογώ πως είναι νομικό το ζήτημα. Αυτή είναι η άποψη που έχει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα τον λόγο έχει η κυρία Γκρέσλε. Και μετά η κυρία Γελασέντερ θα τελειώσει τη συζήτηση. Κοιτάξτε, ε, επειδή βλέπω πως ανοίγουμε και κλείνουμε υπηρεσίες εδώ πέρα. Δεν έχουμε κλείσει ποτέ υπηρεσία. Πλην αυτής που είχε εργαστεί στα Βαλκάνια και ήταν εκτελεστική της Κομισιόν. Αλλιώς δεν έχει κλείσει ποτέ η υπηρεσία. Έχουμε 37 αυτή τη στιγμή. Ενώ πριν από λίγα χρόνια είχαμε μόλις τέσσερις τέτοιες υπηρεσίες. Οπότε... Εάν ε, κλείσει αυτή η υπηρεσία, και πάνε οι αρμοδιότητες της ΣΕΠΟΛ. Δεν ξέρω, να βρίσκω λίγο υπερβολικό και πραγματικά θα ήθελα να μάθω τι, τι παίζεται σε αυτό το φάκελο. Προξενεί πραγματικά έκπληξη. Και δεν ξέρω γιατί υπάρχει το συναισθηματισμός. Πρέπει να μπορούν να γίνουν πράγματα τα οποία είναι λογικά. Με τη Γιούτα Χάουκ ήμασταν μαζί στην ομάδα εργασίας και πάνω από ένα χρόνο το συζητούσαμε, το παρουσιάσαμε τα συμπεράσματά μας στην Ολομέλεια, ψηφίστηκε και ξαφνικά ε, όλοι κάνουν πίσω. Δηλαδή να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Θεωρώ πως κάποιο λάθος κάνουμε. Οι δε υπηρεσίες αυτές που εντωμεταξύ έχουν γίνει 37, όλοι οι πολίτες θεωρούν πως είναι υπερβολικά πολλές. Και φτάσουμε σε 50 τον αριθμό και θα έχουμε ένα τεράστιο μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα γίνει χωρίς εμάς. Κλασικά μέσα του Συμβουλίου αυτά. Προσπαθήσαμε λίγο να εκδημοκρατήσουμε την ε, κοινή αυτή προσέγγιση. Να, δεν ξέρω. Η καημένη Γιούτα δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. δεν ξέρω γιατί συζητάμε τέτοια ζητήματα και μετά όταν φτάνει η στιγμή λέμε «Ε, μα δεν το θέμα όμως τελικά να γίνει κάτι τέτοιο». Ο Ιωλασέντερ και η Bueno, seguramente yo me explico mal porque. Eh, Προφανώ δεν τα λέω καλά. Es muy joven. Es decir, yo como soy más vieja que ella. Είναι και νέα η κυρία Γκρέσλε. Εγώ είμαι πιο γριά και έχω πολλά χρόνια εδώ. Δούλευα και στην Γραμματεία πριν γίνω βουλευτής. Μπορείτε να ρωτήσετε, να δείτε στον τύπο τι είχε γίνει με όλα αυτά τα μπάτς, ε, το Λεωνάρντο. Η αρχή της ανάθεσης στο εξωτερικό καθηκόντων που δεν μπορούσε να ελοποιήσει η ε, επιτροπή έπαιρνε του κόσμου τους ειδικού, προσωπικό έκτακτο κλπ. Μετά την υπόθεση Σαντέρ άλλαξε η κατάσταση. Εγώ μιλώ για αυτές που δημιουργήθηκαν μετά. Τις ε, υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν μετά. Διότι 37 υπηρεσίες έχουμε, 28 κράτη-μέλη, όταν του εξηγούμε πράγματα τα καταλαβαίνει. Υπάρχουν κράτη-μέλη που είναι ευχαριστημένα, πανευτυχοί που έχουν γραφεία στο εδαφό του. Δουλεύουν με τους οργανισμούς αυτούς και φροντίζουν να είναι πιο αποτελεσματικά. αποτελεσματικά. Εμείς τα ψηφίσαμε άλλαστε, η Ολομέλεια τα ψήφισε. Μπορεί να υπάρχουν αντιπαραθέσεις, αλλά νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να δουλεύουν καλά οι υπηρεσίες αυτές. Όσο περισσότερο μπλέκουμε τα πράγματα, όσο περισσότερα καθήκοντα επιβάλλουμε, τόσο ευκολότερα, τόσο δυσκολότερος γίνεται ο έλεγχος. Μία διαδικασία που είναι ξεκάθαρη και ε, ε, ασκεί η Europol τα καθήκοντα που της λέει η συνθήκη. Έρχεται ο εκπρόσωπος της και μου λέει δεν το απαγορεύει η συνθήκη. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Ότι επειδή δεν το αναφέρει σημαίνει πρέπει να το κάνει. Το ότι δεν εμφανίζεται δεν σημαίνει ότι επεκτείνεται η αρμοδιότητά της. Το ότι το λέει αυτό η Βρετανική, το Βρετανικό δίκαιο δεν σημαίνει ότι συμβαίνει πάντα. Οι συνάδελφοι που δουλεύουν κάθε μέρα με την Europol το ξέρουν. Όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα αστυνόμευσης στην Ευρώπη μας λένε ότι η Europol πρέπει να μείνει ως έχει και η ΣΥΠΟΛ ως έχει. Το να φέρουμε τη ΣΥΠΟΛ στη Χάγη άσχημα δεν νομίζω ότι θα διευκολύνουμε την ελεγκτική ικανότητα του Κοινοβουλίου. Εγώ θα ζητούσα να υποστηρίξετε τις θέσεις με το συντομότερο δυνατό για να κρατήσουμε τη σαφήνεια, τον ειδικό χαρακτήρα κάθε υπηρεσίας και την ικανότητα του Κοινοβουλίου να ολοκληρώνει τον έλεγχο που απαιτείται και της Επιτροπής να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα. Αυτά και ευχαριστώ. Köszönöm Με αυτά κλείνουμε την ημερήσια διάταξη. Επόμενο θέμα, το σημείο 12. Τροποποίηση του κανονισμού 9 12 για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού GNSS. Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού. Και εδώ είναι η υπεύθυνη κυρία Γιάλα Σέντερ. Παρακαλώ κυρία Γιάλα Σέντερ. Ξανά ευχαριστώ. Πρόκειται για τον οργανισμό GNSS, το παλιό Γαλιλαίο. Εδώ προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ικανότητα του οργανισμού αυτού να αντιμετωπίσει τις νέες ε, αποστολές που έχει αναλάβει. Την αποστολή και τον έλεγχο στον προπολογισμό της υπηρεσίας αυτάς. Οι τροπολογίες μου είχαν στόχο να θέσουν έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση τη στιγμή της εκλογής του, του εκτελεστικού διευθυντή του οργανισμού. Εμεί ακολουθούμε δηλαδή το ίδιο μοντέλο και σε άλλους οργανισμούς που διαθέτουν διευθυντή θέλουμε να μπορούμε να διατηρήσουμε ισχυρό το ρόλο του Κοινοβουλίου εκεί, ούτως ώστε πριν τον ορισμό την τοποθέτηση του Διευθυντή να υποβάλλεται σε ακρόαση από το Κοινοβούλιο. Επίσης ανασφάρομαι στην, στην ανάγκη να υπάρξει διαχωρισμός. Η Επιτροπή έκανε μια βαθιά μελέτη των εναλλακτικών λύσεων για το θέμα των διαφορετικών καθηκόντων της παλιάς και της νέας επιχειρησιακής αρμοδιότητας του οργανισμού αυτού. Τόνισε λοιπόν την ανάγκη να τεθεί την πρώτη, ε, από, την πρώτη στιγμή και αυτό μας το λέει η Επιτροπή και έχω δουλέψει στην Επιτροπή για το Γαλιλαίο με όλα τα προβλήματα που είχε καταλαβαίνω ότι σε αυτή, την πρώτη, η πρώτη στιγμή είναι μια αυτή η πρώτη απόφαση είναι καλή απόφαση. Ο διαχωρισμός των δύο τομέων δράσης του οργανισμού για να αποφευχθούν συγκρούσεις συμφερόντων. Ενίσχυσα με τις τροπολογίες μου το άρθρο που έχει να κάνει με τη σύγκρουση συμφερόντων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οργανισμός αυτός, όπως και η ΕΑΣΑ, ο Οργανισμός Ασφάλειας των Αεροπορικών Μεταφορών, έχει ένα μικρό αριθμό εμπειρογνωμόνων. Βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο κόσμο με μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη και υπάρχουν πολλοί ειδικοί παντού. Ζητώ λοιπόν να υπάρξει καλύτερη διαχείριση και έλεγχος των συγκρούσεων συμφερόντων. Καταλαβαίνοντας ωστόσο και από την άλλη ότι δεν φυτρώνουν στα δέντρα οι μηχανικοί. θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν και καλοί εργαζόμενοι στις υπηρεσίες. Πιστεύω ότι με τις τοπολογίες βελτιώσαμε τα κείμενα. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. η Επιτροπή, επειδή χρειάστηκε να αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις την ικανότητα του οργανισμού αυτού να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις, έχει κάνει μια αποδεκτή πρόταση. Είμαι έτοιμη να ακούσω τις προτάσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Καβαντά ζήτησε το λόγο. Μιστέρ ε, Σνίτγκερ. Όχι, με συγχωρείτε. Ο κύριος το έχει το λόγο. Άλλο όνομα είχα εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι η κυρία Καβαντά δεν μπόρεσε να έρθει. Ευχαριστώ και την κυρία Καβαντά. Η κυρία Γιάλα Σέντερ τόνισε στην εισαγωγή της τις λόγους για την πρόταση αυτή. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τρομοποιήσουμε, να εφαρμόσουμε ε, αυτό το οποίο έχει προκύψει ως συνένεση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τα δύο προγράμματα Τζίνεσες Γαλιλαίο και Έγνος. Και βασικό στοιχείο είναι ο αυξημένος ρόλος της ε, υπηρεσίας αρμόδιας για το GNSS της λεγόμενης GSA που όπως ξέρετε βρίσκεται στην Πράγα. Στόχος και πρόθεση είναι να δώσουμε ένα μεγαλύτερο ρόλο στην επιχειρησιακή λειτουργία του Γαλιλαίου και του Έγνος και βεβαίως αυτό πρέπει να αντισταθμιστεί με επιπρόσθετα μέτρα για να καθορίσουμε το συγκεκριμένο αυτό κομμάτι που είναι βεβαίως ε, πιστοποίηση ασφάλειας. Το είπε πολλές φορές η κυρία Γιάννα Σέντερ. Όντε βέβαια δηλαδή να υπάρχουν συγκρούμενα συμφέροντα. Υπάρχουν λοιπόν εδώ πέρα δύο τομείς αρμοδιοτήτων ευθύνης που πρέπει να είναι διακριτή αφενός υπάρχει τρέχουσα ευθύνη για την πιστοποίηση ασφαλείας αφετέρου κάτι το οποίο θα γίνει από το 2014, η αυξημένη επιχειρησιακή ευθύνη για τα συστήματα, γιατί πρέπει να τα διαχωρίσουμε αυτά. Είναι απλή απάντηση. Εάν ε, υφίσταται κανείς πίεση για να εκτοξεύσει δορυφόρο, τότε μπορεί να θέλει κανείς να ελέγξει τις αποφάσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να αναβάλουν μια τέτοια εκτόξευση. Γι' αυτό η Κομισιόν θεωρεί πως πρέπει να ενισχύσουμε το λεγόμενο συνικό τείχος μεταξύ των δύο αυτών λειτουργιών. Τρία μέτρα έχουν προταθεί. Το ένα αφορά την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας. Έχουμε αφενός την ευθύνη του δοσού να επεξεργαστεί το πρόγραμμα εργασίας. Από την άλλη υπάρχει το λεγόμενο Συμβούλιο Πιστοποίησης Ασφαλείας. Δεύτερον, το ίδιο ισχύει και για τις εκθέσεις, οπότε η αρμοδιότητα του εκτελεστικού διευθυντή ε, που είναι να αναφέρει στην Κομισιόν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας και βεβαίως ο πρόεδρος του Συμβουλίου Πιστοποίησης Ασφαλείας που θα δίνει και αυτός λόγο. Και το τρίτο κομμάτι του συνοικού αυτού τείχους αφορά το προσωπικό όπου προτείνει η Κομισιόν να δοθούν περαιτέρω αρμοδιότητες στον πρόεδρο του Συμβουλίου Πιστοποίησης Ασφαλείας για τυχόν κυρώσεις. Αυτός είναι ο βασικός στόχος της πρότασης αυτής. Δηλαδή να ευθυγραμμίσουμε τον κανονισμό με αυτά τα οποία έχουν προκύψει ε, ως συνένεση για τη διακυβέρνηση του προγράμματος. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε είναι η ευθυγράμμιση του κειμένου με την κοινή προσέγγιση, οπότε Απλά προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αλλαγές οι οποίες θα ισχύσουν σε όλες τις νομικές βάσεις ε, και βεβαίως θα πρέπει να δώσουμε και τους απαραίτητους πόρους για να μπορείς να λάβει τις νέες ευθύνες η υπηρεσία αυτή. Σε σχέση με αυτό λοιπόν και το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Αγιά Σέντερ, Συμφωνούμε πλήρως με την πρόθεση του Κοινοβουλίου να αυξηθεί η λογοδοσία και η διαφάνεια, να μην υπάρχουν συγκρόμενα συμφέροντα και θα εξετάσουμε στενά τις προτάσεις της κυρίας Αγιάλα Σέντερ για την αναδιατύπωση μιας ε, ή κάποιας άλλης ευτυχής, αλλά επί της αρχής δεν έχουμε σοβαρές διαφωνίες. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητάει το λόγο. Κυρία Γιάλα Σέντερ, θέλει να πει κάτι άλλο. Έχετε το λόγο. Τίποτα να ευχαριστήσω την επιτροπή του συναδέλφου. Τεχνικό είναι το θέμα βέβαια, αλλά αν υπάρχουν άλλες τοπολογίες είμαι στη διάθεσή σας.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 Είχα ξεχάσει να σας αγγείλω κάτι και συγγνώμη. Στο προηγούμενο σημείο το Σίπολ και Europol και την πιθανή συγχώνευση η προθεσμία υποβολής των υπολογιών είναι 18 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, αύριο δηλαδή. Το ίδιο, την ίδια προθεσμία, έχει και το θέμα που τώρα συζητήσαμε. Το GNSS. Πάλι δηλαδή 18, 9 του 12 το μεσημέρι. Κυρίε και κύριοι, προχωράμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η ειδική έκθεση 22 του 2012 έχετε δύο έγγραφα. Ειδική έκθεση 22-2012 του Ελεκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Συμβολή στην αποτελεσματική χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων στην ένταξη πολιτών τρίτων χωρών» Ερωτηματικό. Ο κ. Μαρινέσκου έχει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Μαρινέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ισορροπημένη είναι η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, ε, εκτελεστικού συνεδρίου, λαμβάνει ε, υπόψη ε, όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει σε αυτό το πρόγραμμα. Η εργοπορημένη έγκριση της νομοθεσίας, η έλλειψη στόχων και δικτών σε επίπεδο κρατών μελών, ε, οδήγησαν ε, σε παρεμπόδιση των στόχων, στην επίτευξη των στόχων. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο υποδιαπραγμάτευση προτάσεις της Κομισιόν ε, που προτείνουν και νέα δομή αλλά και βελτιωμένη νομοθετική μορφή που θα διευκολύνουν και θα ρυθμίσουν καλύτερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Χωρών και Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες. Στις νέες ε, διατάξεις λοιπόν υπάρχουν ε, ε, κάποιες καλές διατάξεις. Ορισμένα από τα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν είναι η δημιουργία κοινών υποχρεωτικών παραμέτρων των κρατών μελών για την περίοδο 14-15 και δέσμευση των κρατών μελών ότι θα δημιουργήσουν και σε εθνικό επίπεδο αντίστοιχες παραμέτρους. Ε, στη νέα προγραμματική περίοδο 14-20 ε, να μην υπάρξουν πλέον πιστοποιητικές αρχές και απλούστευση ε, των ελέγχων. Αυτά είναι ε, απαραίτητα. Επίσης, δίκτυο ε, διακρύβωσης ε, έτσι ώστε οι βέλτιστες πρακτικές καθώς επίσης και η αξιολόγηση και η επιθεώρηση να γίνονται πιο εύκολα. Ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα στην έκθεση του ελληνικού Συνεδρίου αναφέρεται στις ε, προτεραιότητες όσον αφορά αυτά τα δύο ταμεία για την ένταξη των επικών τρίτων χωρών. Ε, η Κομισιόν προτείνει μεγαλύτερο βαθμό συμπληρωματικότητας μεταξύ των δύο ταμείων και επομένως αυξημένη συνεργασία. Πιστεύω ότι αυτό είναι σωστό να γίνει και ευθυγραμμίζεται και με την αρχή της επικουρικότητας, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη τα οποία επιθυμούν ε, να έχουν την δυνατότητα σε εθνικά ε, προγράμματα να δημιουργήσουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες ε, για, τα, τα, για τα δραστηριότητες που καλύπτουν τα ταμεία αυτά ε, και επίσης και στις εταιρικέ σχέσεις με τα κράτη-μέλη να υπάρχει προωθημένη συνεργασία όσον αφορά τα δύο αυτά ταμεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ λέει ο Πρόεδρος. Τον λόγο έχει ο Μίλεν Μάρτιν Τσβίγκελ, ε, εκπρόσωπος ε, του ελεγκτικού συνεδρίου, να μας πει δύο λόγια όσον αφορά την ειδική αυτή έκθεση. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε σήμερα εδώ. Η βοήθεια προς τους ανθρώπους που έρχονται από τρίτες χώρες ή από χώρες με προβλήματα να ενταχθούν στην κοινωνία είναι πολύ ψηλά στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και βεβαίως κατά αυτήν την έννοια έχουν διευρυνθεί οι δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τη δημιουργία και των ταμείων ε, ένταξη υπηκόντρων των χωρών και ταμείο για τους πρόσφυγες. Προσπαθήσαμε να δούμε εάν πραγματικά βοηθούν τα ταμεία αυτά αποτελεσματικά στην ένταξη των υπηκών τριτών χωρών. Θα πω δύο λόγια για τα ευρήματα και μετά κάποια συμπεράσματα. τα ευρήματα ε, που προέκυψαν ε, από τις εργασίες του ελεκτικού συνεδρίου είναι ότι τα θετικά αποτελέσματα μπορεί να υπάρχουν σε τοπικό μονομένο επίπεδο, αλλά ε, δεν υπάρχει σωστή στοχοθέτηση από πλευράς των ε, κρατών μελών. Επίσης, έγινε μια ενδιάμεση έκθεση από την Κομισιόν που θα έπρεπε να καλύπτει τα αποτελέσματα, αλλά που δεν δίνει όμως αρκετά ε, πληροφοριακά στοιχεία έτσι ώστε να γίνει η σωστή αξιολόγηση. Ούτε Ούτε Κομισιόν, ούτε τα κράτη-μέλη επίσης έχουν αρκετές πληροφορίες για τον ακριβή τρόπο δαπάνης των κονδυλίων. Όσον αφορά το ίδιο το... Τώρα που το MFF τελείωσε όσον αφορά το ίδιο το πρόγραμμα, πρέπει να πούμε ότι μακρά λυσίδα ελέγχων που γίνονται από τις αρχές στα κράτη-μέλη έχει θέσει ένα εξαιρετικά υψηλό διοικητικό άχθος στην όλη διαδικασία. Όλες οι αρχές, όπως και η ίδια η Κομισιόν, έχουν πληγεί από αυτό το βάρος. Ε, βρήκαμε ότι υπάρχουν δυσλειτουργίες ε, παρά τις ε, ε, τα εχέγγυα τα οποία εξ αρχής είχαν μπει στο πρόγραμμα. Ε, από εκεί λοιπόν, από τις λειτουργίες αυτές προκύπτουν καθυστερήσεις όσον αφορά τα αρχικά προγράμματα, όσον αφορά ε, τα επιπλέον προγράμματα ελλειπή καθοδήγηση, έλλειψη κατανόησης όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των τριών αρχών. Ε, υπήρξαν ε, αδυναμίες ε, και στον τρόπο διαχείρισης των ελέγχων που δεν έγιναν σε αρκετά πρώιμο στάδιο από την Κομισιόν και που επομένως προκάλεσαν προβλήματα από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Επίσης βρήκαμε ότι αυτά τα προβλήματα ε, τελικά μείωσαν ε, το, την αποτελεσματικότητα ή και την ίδια την ε, δυνατότητα ολοκλήρωσης των προγραμμάτων. Είχαμε μονάχα 66% ολοκλήρωση για το, 2007, συγγνώμη, για το 2012 και λίγο παραπάνω για το 2013. Όπως ε, είπε και ο ίδιος ο κύριος Μαρινέσκου και όπως γνωρίζετε, η Κομισιόν ε, έχει ήδη αντιδράσει στα πλαίσια και του πολιετούς δημοσιονομικού ε, προγράμματος, κάνοντας κάποιες νέες προτάσεις, οι οποίες αφορούν μονάχα την περίοδο 14-20. Βάσει του οικονομικού μας ελέγχου, στην ε, συγκεκριμένη περίπτωση εμείς ελέγξαμε ε, και το επερχόμενο πολιετές πρόγραμμα και μέσω επιστολής τον Ιούλιο του 2012 είχαμε εκφράσει άποψη όσον αφορά τις προτάσεις, τις νέες προτάσεις της Κομισιόν. Ωστόσο, μία από τις συστάσεις μας και που ε, παραμένει ακόμα ανεκπλήρωτη στην, ε, ε, ε, εμείς καταλήξαμε σε έλλειψη συντονισμού με άλλα ευρωπαϊκά ταμεία και χαμηλό βαθμό αποτελεσματικότητας. Επίσης, καταδεικνύεται βάσει, της οικονομικής, βάσει του οικονομικού ελέγχου ότι τα περισσότερα μέτρα θα μπορούσαν να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ας πούμε μαθήματα γλωσσικά για υπηκόους τρίτων χωρών ε, από το, χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Ταμείο Ένταξη Υπηκών Τρίτων Χωρών, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων. Δηλαδή τρεις, τρία διαφορετικά ταμεία, ε, τρία, τρεις ε, πόροι που πληρώνουν, τρία στα τρία λεωφορεία που να πληρώνουν εισιτήριο για το ίδιο πράγμα. Κάτι γίνεται λοιπόν, δεν λειτουργεί καλά το σύστημα. Γι' αυτό ακριβώς ε, στην έκθεσή μας ε, ε, ζητούμε συνολική αξιολόγηση που πρέπει να γίνει άσχετα εάν οι μετανάστες προέρχονται από τρίτες χώρες ή από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρξει και μια σωστά σχεδιασμένη χρηματοδοτική μορφή, χρηματοδοτικό εργαλείο καλά σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Επομένως, τους ιώδες πρόβλημα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξη Υπηκόντρων των Χωρών σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί. Χαίρομαι που στην πρόταση του κυρίου ε, Μαρινέσκου δίνεται και μια άλλη δυνατότητα έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δύο ταμεία, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκών τρίτων χωρών ε, κατά κάποιο τρόπο να συγχωνευτούν. Ε, στην τελευταία παράγραφο της ε, προτάσεως λαμβάνεται υπόψη η αρχή της επικουρικότητας έτσι ώστε να δοθεί στα κράτη-μέλη τα οποία επιθυμούν να προβλέψουν στα εθνικά τους προγράμματα ε, την δημιουργία περαιτέρω συνεργειών για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, διασφαλίζοντας ότι και στις ε, συμφωνίες εταιρικέ ε, σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών ενδυναμώνεται το σκέλος αυτό. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν όχι μόνο η προκείμενη έκθεση αλλά και άλλες εκθέσεις ευθυγραμμίζονται με τα ευρήματα που προέκυψαν από τον δικό μας οικονομικό λογιστικό έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο Μάρτιν Σίφερ και η Σένσου Μακοβέη. Δεν ξέρω αν κάποιο θέλει να πάρει το λόγο εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α, ποιος από τους δύο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Έχουμε ήδη εκφράσει τις απόψεις Κομισιόν επί των συστάσεων που έκανε το Ελληνικό Συνέδριο και καλωσορίζουμε και το έγγραφο του εισηγητή επί της εκθέσεως του Ελληνικτικού Συνεδρίου. Καθώς θεωρούμε πως όλα πηγαίνουν προς την σωστή κατεύθυνση και συμφωνούμε με τις περισσότερες συστάσεις του συνεδρίου και πολλά από τα πράγματα που τονίζει ο κύριος Μαρινέσκου καθώς όπως ξέρετε είναι και εισηγητής για ένα από τα νέα χρηματοδοτικά μέσα στον τομέα των εσωτερικών, το μέσο για την ε, εσωτερική ασφαλεία των συνόρων. Ε, ήδη έχουμε πει επανειλημμένως πως... Ε, ε, Υιοθετήσαμε πολλές από τις ε, συστάσεις που αναφέρονται στο έγγραφο εργασίας και βεβαίως αυτό θα το δείτε και στο έγγραφο εργασίας πολλά πράγματα τα έχουμε αντιμετωπίσει όσον αφορά την απλοποίηση πέρασαμε σε, μια, σε ένα πολιετή προγραμματισμό αυξήσαμε την διαφάνεια μέσω της ε, υποχρεωτικής ε, εταιρική σχέσης με πλήρη διαφάνεια και καταργήσαμε μία από τις τρεις αρχές που εμπλέκονται αυτή τη στιγμή σε εθνικό επίπεδο με τη διαχείριση των κονδυλίων οπότε υπάρχει μόνο η ελεγκτική αρχή και η αρμόδια αρχή δύο μόνο αρχές στο εθνικό επίπεδο και Βεβαίω, δεν γίνεται κάποια διάκριση στο μέλλον μεταξύ των τεσσάρων διαφορετικών μέσων στο τομέα των μεταναστευτικών, δηλαδή σύνορα, επιστροφές, ε, πρόσφυγες ε, και τα λοιπά. Τρία από αυτά λοιπόν τα ταμεία θα ενσωματωθούν στο ένα ενιαίο ταμείο ασύλου και μετανάστευση και απλοποίηση αυτή θα οδηγήσει σε μια πιο αποτελεσματική διαχείριση του Ταμείου. Επίσης έγιναν κάποιες συστάσεις σε σχέση με τη συμπληρωματικότητα με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το γνωρίζουμε, αλλά έχουμε πει επανειλημμένως πως Πέρα από αυτή τη συμπληρωματικότητα, η διασφάλιση αυτή είναι βασικά έργο των αρχών στο εθνικό επίπεδο. Δυστυχώς οι αρμόδιες αρχές είναι διαφορετικές σε κάθε χώρα, οπότε δεν είναι εύκολο για τα κράτη-μέλη να παρακολουθήσουν την κατάσταση. ιδέως παραμένει κυρίως αρμοδιότητα των κρατών δεύτερων θέλω να πολιτική και από νομική σκοπιά. Τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το κοινωνικό ταμείο και τα ζητήματα ολοκλήρωσης που αντιμετωπίζει το μελλοντικό αυτό ταμείο ασύλου και μετανάστευσης, το τωρινό ενσωμάτωσης, ε, δεν αντιμετωπίζουν τα ζητήματα σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Είναι η διαφορά μεταξύ ένταξης για λόγους κοινωνικής ένταξης ή αν είναι μέρος μιας κοινή μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα. Αν δούμε την δύσκολη συχνά διάκριση μεταξύ δράσεων που αφορούν μέτρα κοινωνικής ένταξης και αφορούν τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι σαφές, έτσι, οι υπήκοοι της Ένωσης δεν ε, είναι δυνατόν να είναι αντικείμενα μέτρων ένταξης γιατί έτσι περιορίζουμε την ε, ελευθερία μετακίνησης που έχουμε. Είναι ξεκάθαρα τα όρια. Οπότε το Ταμείο Ένταξης δεν μπορεί να συμπεριλάβει υπηκόους Ένωσης. Όμως, στο νέο μέσο, αν δείτε την πρόταση της Κομισιόν, το άρθρο 9, ε, συμπεριλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο ρεαλισμό. Και προσπαθήσαμε να δούμε και τα εφαρμοστικά μέτρα για τις ΜΚΟ και τις ε, αρχές οι οποίες εφαρμόζουν τα μέτρα συμπεριλαμβάνοντας και άτομα με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή έργων που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν από το πεδίο εφαρμογής του μελλοντικού αυτού ταμείου. για να στηρίξουμε ένα έργο που απευθύνεται κυρίως σε υπηκόρους τρίτων χωρών. Μέχρι εκεί πάμε και το βλέπετε αυτό και από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και στην ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Βλέπετε πως Το θέμα αυτό λοιπόν είναι διχαστικό, κάποια κράτη-μέλη ε, συμφωνούν περισσότερο με την Κομισιόν, κάποια άλλα α, ε, ακολουθούν μια πιο νομική προσέγγιση και λένε πως είναι κάτι το θεμελιώδες που πρέπει να γίνει σεβαστό και ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε μέτρα ένταξης για υπηκόσους ένωσης. Πότε περιοριστήκαμε Βρισκόμαστε σε μια λύση που είναι σε ευριακό στάδιο αυτή τη στιγμή. Και αυτά έχω να πω μέχρι στιγμής για τις ε, παρατηρήσεις του εισηγητή. Και του ελεκτικού συνεδρίου. Λαμβάνοντα υπόψη λοιπόν όλες αυτές τις παρατηρήσεις, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις τριμερεί με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, οπότε το να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες ίσως να μην είναι απολύτως σωστό όπως είπα εκρεμεί ακόμα ο, ο διάλογος. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ερωτώ. Θέλει κάποιον λόγο. Δεν βλέπω. Κάποιον να ζητάει το λόγο. Από ό,τι φαίνεται. Είχαμε μια πολύ καλή πρόταση ε, του κ. Μανέσκου και άρα του δίνω πάλι το λόγο. Thank you very much. Just... Uh, Ευχαριστώ πολύ. Μια παρατήρηση προς την Επιτροπή. Είναι γεγονός, αληθεύει ότι αυτή τη στιγμή γίνονται διαπραγματεύσεις όσον αφορά ε, τα ταμεία αλλά βλέπω ότι η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη ε, τις εξελίξεις ε, και, λαμβάνει, και, και συμπεριλαμβάνει μάλλον και όλα τα μεμονωμένα στοιχεία της συμφωνίας αλλά λαμβάνει υπόψη της όλα αυτά στα πλαίσια και της ε, Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης που αναθεωρείται κάθε τόσο. Διότι ταυτόχρονα γίνονται και διαπραγματεύσεις ε, ανάμεσα στις χώρες μέλη και την Κομισιόν για την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης. Να ζητήσω λοιπόν από την Κομισιόν ε, ε, να δει το ενδεχόμενο συμπερίληψης αυτής της σύστασης την επόμενη φορά. Να προσπαθήσουμε δηλαδή τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν όσο γίνεται περισσότερη συνέργεια μεταξύ των ταμείων. Τώρα ξέρετε ότι επιτρέπεται να χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα από περισσότερο από ένα ταμεία ε, κοινωνικό, συνοχής, ε, περιφερειακή ανάπτυξης κτλ. Αν είναι δυνατόν λοιπόν να αξιολογηθεί αυτή η δυνατότητα, η οποία θεωρώ ότι θα αποβεί προς όφελος ε, μιας καλής διαχείρισης δαπανών. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι κλείσαμε το σημείο αυτό στη μέση διάταξη. Δεν έχω κάτι για τα διάφορα. Κατά συνέπεια, το αφήνουμε και αυτό. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει 25 Σεπτεμβρίου, εδώ, Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ και συμμετάσχετε στη συζήτηση. Πέρα συνεδρίασης.